we Αρχίζουμε λίγο αργά, νομίζω ότι είναι τρεις και τέταρτο. Ελπίζω να είχατε καλές διακοπές του Πάσχα και να είστε έτοιμοι για εργασία τώρα. Ε, έχουμε εδώ στην άλλη Δευτέρα, η Πρωτομαγιά είναι αργία, οπότε και πάλι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μια μικρότερη εβδομάδα. Μου λέχθηκε ότι ο κύριος Σκούλογλου δεν μπορεί να είναι εδώ για το σημείο 15 και συνεπώς ε, θα έχουμε ε, μόνο την συζήτηση ανθρώπινα δικαιώματα τρίτων χωρών. Θα έχουμε λοιπόν μια σύντομη συζήτηση πρωτού ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση, αλλά κρατάμε την προθεσμία για τα μέλη που είναι 3 Μαΐου για τις τροπολογίες. Ε, στις 6 ε, το απόγευμα, 3 Μαΐου, είναι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Αυτή είναι η μόνη αλλαγή που έχω. Μπορούμε να υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη. Απλώς μία αναγγελία την Τετάρτη η ε, Επιτροπή μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει ειδική εκδήλωση την ε, Πέμπτη, την Τετάρτη θα συζητήσουμε ε, την εισήγηση στην Ολομέλεια και ε, θα ε, έχουμε ναι, την, ε, την επέτειο για την καταστροφή που έγινε τότε για την επίθεση στην, στην αίθουσα 5G3. Θα δείτε λοιπόν την πρωτοβουλία Γκάρμαν και θα έχουμε την οργάνωση που εκπροσωπεί το δίκαιο, ηθικό εμπόριο και θα μιλήσουν για τη δική τους πρωτοβουλία δεν έχουμε εδώ τώρα πολλούς συναδέλφους, θα στείλουμε μια υπενθύμηση στο τέλος της ημέρας, διότι μετά την, ε, τις διακοπές δεν ξέρω αν θα έρθουν πολλοί να εργαστούν. Έχουμε τώρα το σημείο 3, έχουμε την, ε, ε, την, ε, τα πρακτικά της 28ης Φεβρουαρίου. Βλέπω ότι δεν έχουμε παρατηρήσεις και αυτό έχουμε το 4 υιοθέτηση των αποφάσεων και συστάσεων των συντονιστών αν έχετε παρατηρήσει στη γραμματεία μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Αν δεν έχουμε καμία παρατήρηση θα θεωρήσω ότι τα πρακτικά αυτά έχουν υιοθετηθεί. Έχουμε τις αναγγελίες από την Επιτροπή στο σημείο 5. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Στις 3 Μαΐου η Επιτροπή ε, και είπα ότι εκπρόσωπος θα αναφέρουν την κοινή ανακοίνωση ε, για την εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής, ούτως ώστε όλοι να ξέρετε και το περιεχόμενο είναι η προετοιμασία των στρατηγικών ε, στόχων για την διάσκεψη του Νοεμβρίου και θα δώσουμε για μια νέα όθηση που θα ανταποκρίνεται στις αλλαγές ε, των εποχών μας, ε, το νέο θεματολόγιο 2030 και νομίζω ότι η ΕΦΚΟ επίσης ε, θα θέλει να συμμετάσχει και να παρουσιάσει την ανακοίνωση και να συζητήσει αλλαγές που θα θέλατε να επιφέρετε. Ευχαριστώ βεβαίως. Θέλουμε να έχουμε μια παρουσίαση από την Επιτροπή μας. Συμφωνήσαμε να πάρουμε άδεια για, για, την μια γνωμοδότηση για την Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Πρόκειται για ένα θέμα κλειδί για την δική μας Επιτροπή. Θα έχουμε λοιπόν διάλογο μαζί σας και θα προσπαθήσουμε να βρούμε χρόνο για να έχουμε τον ε, Επίτροπο και την ύπατη εκπρόσωπο για μια παρουσίαση για την στρατηγική. Αργότερα σήμερα θα το κάνουμε αυτό σύντομα. Βεβαίως έρχεται ο Μάιος πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Σημείο 6. Η Έλλη Σλάιν είναι καθοδόν και θα έρθει από μια μια στιγμή στην άλλη ούτε είναι εδώ. Μήπως ξέρετε, ξέρει το προσωπικό αν είναι καθοδόν. Θα περιμένουμε λοιπόν για το σημείο 6, για την Ellie Schlein. Σήμερα είναι μέχρι τις 5.30, μέχρι τις 5.30 που έχουμε την ψηφοφορία την ψηφοφορία για το, με την ΑΦΕΤ και την Επιτροπή Προϋπολογισμού στην αίθουσα 3C50. Εδώ σε αυτό το κτίριο είναι σημαντικό να έχουμε αρκετά άτομα εκεί για αυτήν την ψηφοφορία για την, στο, την φάκελο της συναπόφασης. Θα έχουμε λοιπόν αυτό το θέμα στις 5.30 στην άλλη αίθουσα να τονίσω το ίδιο με εσάς, γιατί είμαστε σε μικρή επιτροπή και πρέπει να είμαστε παρόντες για να μπορέσουμε να περασπιστούμε την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Ακριβώς. Θα γίνει η ψηφοφορία και ο κύριος Φρουζουλίκα, ο, ο Σιώδης μας, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά μας έχει πει πόσο σημαντικό είναι το θέμα. Θα περιμένουμε δύο λεπτά τώρα για την κυρία Σλάιερ. Υπάρχει πάντα αυτό το πρόβλημα της Δευτέρης, καθώς έχουμε διάφορες πτήσεις. Να πω επίσης στην ομάδα ότι η ιδέα ήταν να ψηφίσουμε σήμερα και να ψηφίσουμε για το θέλουμε να ξεκινήσουν οι τριμερείς διάλογοι. Υπάρχει ε, ανάγκη να έχουμε απαρτία για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για τους τριμερούς. Ελπίζω οι ομάδες ε, στις τρεις επιτροπές να εργάζονται ώστε να έχουμε τα 71 μέλη που χρειάζονται γιατί είναι η άφετη μπάτζετ και η δική μας ε, Επιτροπή ε, και είναι Δευτέρα απόγευμα η ψηφοφορία. Πρέπει δύο φορές να ελέγξουμε αν θα είναι όλοι εκεί, γιατί ε, πρέπει οπωσδήποτε να είναι όλοι. Θα δώσω λίγο χρόνο στην κυρία Σλάιρ να καθίσει για να μπορέσει να μιλήσει. Ε, οπότε κάνω την εισαγωγή στο θέμα. Σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης, ε, για, η δράση για την ε, βιωσιμότητα. Όπως ξέρουν οι συνάδελφοι, ένα χρόνο μετά την ε, δημοσίευση και την έγκριση της Ατζέντα 2030 το περασμένο Νοέμβρη, η Κομισιόν ε, δημοσίευσε ένα πακέτο ε, ανακοινώσεων για το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να, κάνει, ε, να πάει περαιτέρω την ατζέντα. Αυτό το πακέτο έχει ε, μεν το συνένεση, την Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη, αλλά έχει και μία ανακοίνωση για τα επόμενα βήματα για το βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον, για το οποίο είναι ο πρόεδρος Τίμερμανς ε, υπεύθυνο. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, ετοιμάζει μία απάντηση στην ανακοίνωση ο Σεπ είναι ο εισηγητής. Θα έχουμε από το Συμβούλιο επίσης τα συμπεράσματα για την ατζέντα που θα εγκριθούν στις 20 Ιουνίου και έχουμε και εμείς συντάξει μία γνωμοδότηση. Η Έλλη Σλάιρ είναι η εισηγήτρια και έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Η Ατζέντα 2030 είναι μια φιλόδοξη, γενναιόδορη ατζέντα με μεγάλο ε, δυναμικό για μεταβλητότητα και ε, αφορά στόχους που απαιτούν άμεση δράση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικό ρόλο να παίξει στην εφαρμογή της νέας ατζέντα για την ανάπτυξη, αν σκεφτούμε τις τα τρέχοντα γεγονότα. Θα πρέπει να παίξουμε σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, ως τώρα τα σχέδια που έχουμε δεν είναι επαρκή. Πρέπει να τα συμπληρώσουμε με μια κοινή στρατηγική και ένα πλαίσιο εφαρμογής των ευρωπαϊκών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Έτσι τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να διασφαλίσουν το συντονισμό, την καθοδήγηση και να παρακολουθούν την διαδικασία εφαρμογής. Εγώ ζητώ από την πρώτη μέρα μια ισχυρή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλιστα στη Νέα Υόρκη, μετά από την έγκριση της ατζέντα έγινε αυτό. Και καλωσορίζουμε την ανακοίνωση για τα επόμενα βήματα, όμως για να είμαστε ειλικρινείς περιμέναμε περισσότερα. Δυστυχώς η ανακοίνωση δεν έθεσε έναν ξεκάθαρο δικό χάρτη εφαρμογής και δεν έδωσε μια γενικότερη στρατηγική, απλώς ε, συνδύασε υφιστάμενες πρωτοβουλίες. Θέλουμε λοιπόν νέες πρωτοβουλίες σε βάση των κενών που έχουμε διαπιστώσει και να έχουμε εξωτερικές και εξωτερικές πολιτικές οι οποίες θα ευθυγραμμίζονται με τους στόχους και θα σέβονται την αρχή της ανάπτυξης. Μια ολοκληρωμένη και ε, ε, ε, σημαντική ατζέντα είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα πρέπει να έχει λογοδοσία, παρακολούθηση εξέταση, ένα πλαίσιο δηλαδή που θα περιλαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους ενδιαφερόμενους και την κοινωνία των πολιτών. Η εφαρμογή της Ατζέντα 2030 είναι μια μεγάλη οικονομική δέσμευση. Είναι ένα εργαλείο του κεκτημένου, αλλά δεν πρέπει να είναι το μόνο. Η φορολογική δικαιοσύνη και η διαφάνεια είναι επίσης σημαντικά στοιχεία που θα διασφαλίσουν ότι οι δημοσιονομικοί πόροι που είναι διαθέσιμοι θα φτάσουν για την ατζέντα. Επίσης πρέπει να κεμίσουμε το κενό των 2,5-3 ευρώ που απαιτείται για τους στόχους. Θα πρέπει και ο ιδιωτικό τομέας επίσης να παρακολουθείτε για να διασφαλίζουμε ότι βοηθά στους στόχους της ανάπτυξης και ότι ε, μας ε, πηγαίνει προς ε, βιώσιμες μορφές κατανάλωσης στην Ευρώπη και παγκοσμίω. Επίσης, οι εμπορικές πολιτικές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την ατζέντα και να ευθυγραμμίζονται και με τις αλυσίδες αξίας που έχουν να κάνουν με τη δέωσα επιμέλεια των εταιριών ε, και την ε, πλήρη αλυσίδα τροφοδοσίας. Η μετανάστευση επίσης είναι μια παγκόσμια πρόκληση, ζητά, επιζητά κοινή δράση σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να επαναδιατυπώσουμε την προσέγγιση μας και να λάβουμε υπόψη μας τους στόχους, κυρίως το στόχο 10, βάσει μιας αφήγησης για την μετανάστευση και τους πρόσφυγες που θα είναι θετική. Πρέπει να έχουμε ισχυρή πολιτική βούληση για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη μετάβαση προς ένα βιώσιμο μέλλον. Να μην μείνει κανείς πίσω. Είναι σημαντικό αυτή η Επιτροπή να συνεισφέρει σε αυτή την έκθεση σημαντικά και γι' αυτό αδειμονώ να συνεργαστώ με όλους τους συναδέλφους και να δεχτώ τα σχόλιά σας. Thank Ευχαριστούμε πολύ. Όλοι οι σκιώδεις δεν είναι εδώ. Ε, βλέπω όμως κάποιους συναδέλφους. Μου ζητήθηκε να διαβάσω τις ε, παρατηρήσεις ενός συναδέλφου που είναι απόν. Σας ευχαριστώ λοιπόν, συνάδελφοι, ευχαριστώ την κυρία Σλάιν. Σαν σκιώδης του ΕΛΚ θα ήθελα να σας μεταφέρω κάποιες απόψεις της ομάδας μου. Οι στόχοι για την επόμενη χιλιετία που υιοθετήθησαν από τα Ηνωμένα Έθνη έχουν σαν στόχο την εκρίζωση της φτώχειας και τη διασφάλιση της ανάπτυξης είναι μια συνολική απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Έχουν υπάρξει τεράστιες δημογραφικές αλλαγές, κοινωνικές αλλαγές και περιβαλλοντικού τύπου αλλαγές. Ο πληθυσμός της γης αυξάνεται κατά 80 εκατομμύρια κατ' έτος. Το 2050 το 70% του πληθυσμού θα ζει σε αστικές περιοχές 2,4 δις θα προστίθενται στον πληθυσμό μας από το 2015 μέχρι το 2050, υποθέτουμε. Και η Αφρική επίσης θα αυξήσει τον πληθυσμό της συνταρακτικά. Και αυτό δημιουργεί βέβαια πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα στην υποσαχαρική Αφρική. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν ιδιαίτερα τις ε, μεταναστευτικές ροές, ε, οι οποίες δημιουργούνται πολλές φορές λόγω των άσχημων τοπικών συνθήκων. Και θα πρέπει επίσης ε, και να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι βασικό δικαίωμα να μπορεί κανείς να ζει εκεί που γεννήθηκε και το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να τύχει εγγυήσεων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα Ηνωμένα Έθνη. Η αηφόρος γεωργία είναι το βασικό μέσο για την καταπολέμηση της φτώχειας. Τα δύο τρίτα του πληθυσμού στον κόσμο εξαρτώνται από τη γεωργία για την επιβίωσή τους και υπάρχουν πολλές χώρες δυστυχώς υπό ανάπτυξη οι οποίες εξαρτώνται από γεωργικές καλλιέργειες προς εξαγωγή και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε την κάλυψη των αναγκών σε τρόφιμα και την παραγωγικότητα της γεωργικής παραγωγής, ιδιαίτερα στην Αφρική, ιδιαίτερα στον τομέα τον αγροτοβιομηχανικό, ο οποίος είναι κομβικός για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης βράχη πρόθεσμα και μέσο πρόθεσμα. Χάουταλα. Ευχαριστώ την Έλλη Σλάιν για μια πολύ καλή έκθεση. Είπε τα βασικά. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ατζέντα αυτή είναι καθολικού χαρακτήρα και δεν ισχύει μόνο πλέον για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Καλωσορίζω λοιπόν τις προτάσεις που κάνετε, ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα εφαρμογής με συγκεκριμένους στόχους, προθεσμίες και μεθοδολογία και καλύτερο συντονισμός ανάμεσα στα κοινοτικά όργανα και τα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι η πρόταση υπογραμμίζει την ανάγκη να σχεδιάζονται μεταναστευτικές πολιτικές επί τη βάση συγκεκριμένων δεδομένων. Είναι απαραίτητο αυτό, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την μεταναστευτική κρίση. Υπάρχουν προτάσεις που γίνονται, οι οποίες λειτουργούν μόνο μακροπρόθεσμα, και δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα και στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας. Ως εκ τούτου, στο σημείο 4, σωστά υπογραμμίζονται τα μέσα τα οποία είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση της φτώχειας. Το 0,7% του ΑΕΠ τώρα, σωστά υπογραμμίζονται οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να δίδεται στις λεγότερο αναπτυγμένες χώρες, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης και για τη χρηματοδότηση αηφόρων προγραμμάτων. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και το συγκεκριμένο ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αβιώσιμη Ανάπτυξη. Να υπογραμμίσω επίσης την προσπάθεια η οποία έχει γίνει για τους λεγόμενους εναλλακτικούς δείκτες πρόνοιας. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο χρήζει υποστήριξη στα πλαίσια των συναντήσεων της ομάδας των 20. Έγιναν κάποιες πρώτες συζητήσεις, από τότε τίποτα. Στο σημείο 7, όταν αναφερόμεθα στον ρόλο του ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι χρειαζόμαστε ισχυρές αρχές και κανονισμούς για την κατανομή των ευθυνών. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο και γι' αυτό θα δώσω... Α, όχι, με συγχωρείτε. Θα μιλήσω στα φινλανδικά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης ε, εισηγητής για την ομάδα ΝΤΕ και ε, ασχολήθηκα με το θέμα αυτό. Το σχέδιο γνωμοδότησης είναι πολύ καλό, είναι καλή βάση εργασίας εφόσον περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται. Θα ήθελα στη γνωμοδότησή μας να μιλήσουμε επίσης λίγο περισσότερο για ε, την ουσία θα μπορούσαμε ε, να σκεφτούμε το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η Επιτροπή Ανάπτυξης, η Επιτροπή Περιβάλλοντας ασχολείται με τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, αλλά εμείς τι μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας για να προσθέσουμε ένα λιθαράκι ε, στο όλο κτίσμα σε όλο οικοδόμημα. Πρέπει να αναφερθούμε στην φόρα ανάπτυξη στο κοινωνικό επίπεδο, πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προωθήσει την καλή διακυβέρνηση, τη δημοκρατία τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και αλλού, διότι αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην φόρο ανάπτυξη από την πλευρά του περιβάλλοντος. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει μια δίκαιη ανάπτυξη στις διάφορες περιφέρειες. Θα πρέπει επίσης να προωθήσουμε την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, των μικρών πόλεων, εφόσον υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση ανάμεσα στις ζώνες της υπαίθρου ε, και στις αστικές περιοχές. Θα πρέπει να μιλήσουμε για την ανακύκλωση. Ε, το θέμα του φωσφόρου που τίθεται θα πρέπει αυτές οι θρεπτικές ουσίες ε, να ανακτώνται για να χρησιμοποιηθούν στην οικονομία. Ο ρόλος της γεωργίας όπως τόνισε το ΕΛΚ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει εδώ κατά κάποιο τρόπο να επιβραδύνουμε ε, την ανάπτυξη των μεγαπόλεων που έχει άμεση επιρροή πάνω στους ανθρώπους και αυτός είναι ένας τύπος ανάπτυξης που δεν είναι βιώσιμος και αηφόρος και που έχει επιπτώσεις κοινωνικές στην πολιτική λοιπόν της ανάπτυξης. Θα πρέπει να το λάβουμε αυτό, θα πρέπει στην ανάπτυξη την περιφερειακή να υπάρχει μια συνεκτικότητα, θα πρέπει να επιμείνουμε πάνω σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει να υπάρχει μια ε, συνεκτικότητα ανάμεσα σε αυτό ε, που ζητούμε από τους αναπτυξιακούς μας εταίρους και αυτό που κάνουμε στις χώρες μας και να βασιστούμε σε αξίες ε, που είναι αποδεκτές από όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα δίνω τον λόγο στην Επιτροπή Μαρή Ογελή Βρενά von Brüggen. Δύο έχουμε. Ναι, Ε, ονομάζομαι Τίνα Ντελβά, εργάζομαι στην Γενική Γραμματεία της Επιτροπής που είναι υπεύθυνη για την ανακοινώσει ε, για το θεματολόγιο 2030. Ευχαριστώ τους εισηγητές και τα άλλα μέλη που έλαβαν το λόγο για την συμβολή σε αυτή τη γνωμοδότηση και για τις ε, προτάσεις για την ανακοίνωση της Επιτροπής. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η Κομισιό έχει ε, ηγετικό ρόλο, ε, σημαντικό ρόλο για την θεματολόγιο αυτό και θέλει να συνεχίσει με το ρόλο αυτό. Γι' αυτό στην ανακοίνωση του Νοεμβρίου αναφέραμε δύο θέματα. Πρώτον, θέλουμε την, ε, τους στόχους βιώσιμης αηφόρου ανάπτυξης να τους εντάξουμε στις προτεραιότητες της Επιτροπής η ιδέα ότι η βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να είναι κατευθυντήρια αρχή για όλες τις άλλες πολιτικές και να χρησιμοποιήσουμε τα καλύτερα αριθμιστικά εργαλεία για το σκοπό αυτό. Η νέα δομή της Επιτροπής με αντιπρόεδρο έχει αυτή την προσέγγιση για να προωθήσουμε αυτόν τον σκοπό. Ε, πρώτα απ' όλα ε, πώς ε, να αναπτύξουμε την μακροπρόθεσμη θεώρηση και ε, την πολιτική από το 2020 και ο πρόεδρος Γιούνκερ στην αρχή του Μαρτίου ε, ε, παρουσίασε η Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης και αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας διαδικασίας για προβληματισμό για το μέλλον της Ένωσης σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι θα έχουμε συνεργασία στον τομέα αυτό ε, και ένα από τα έγγραφα ε, στη συνέχεια θα μπορεί να ενδιαφέρει την Επιτροπή σας ε, σχετικά με το θέμα της παγκοσμιοποίησης. Ίσως αυτό το έγγραφο σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και επίσης το έγγραφο θα το έχουμε σε δύο-τρεις εβδομάδες, το Μάιο, και ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια συζήτηση με σας. Η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να τονίσει ότι στο το θεματολόγιο 2030 είναι κοινή ευθύνη όλων, όχι μόνο της Κομισιόν στο επίπεδο το ενωσιακό, αλλά επίσης των αρχών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Δεν είναι μόνο οι αρχές που μπορούν να κάνουν ε, την εργασία, όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι επιχειρήσεις, ε, οι ΜΚΟ, όλοι εμπλέκονται και έχουν ρόλο. Γι' αυτό η Κομισιό αποφάσισε ε, να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για τους εμπλεκόμενους, τους ενδιαφερόμενους και σύντομα θα έχουμε την πλατφόρμα αυτή και θα μπορούμε να σας δώσουμε πιο επίσημες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλει να μιλήσει κάποιο άλλο εκ μέρου τη Επιτροπής. Όχι. Ωραία, επιστρέφουμε στην Έλλη Σλάιν. Ευχαριστώ πολύ όλους τους σκιώδεις ε, για τη συνεισφορά τους και την Επιτροπή για την ε, ενδιαφέρουσα πληροφόρηση κυρίως για αυτή την πλατφόρμα με την πολυμερή Έλαβα υπόψη όλα τα σχόλιά σας. Φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε πώς θα προσθέσουμε αυτά τα στοιχεία στο σχέδιο της έκθεσης για να μπορέσουμε να τα επιτύχουμε. Και όπως ανέφερε και ο Πάμπο η Επιτροπή ΕΜΒΗ έχει τη δική της οπτική. Πρέπει και εμείς να δείξουμε τη δική μας οπτική, να αντικατοπτρίζεται στη γνωμοδότηση, ώστε να είναι πιο ισορροπημένη η ε, προοπτική μας από άποψη ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ. Η προθεσμία είναι 3 Μαΐου το μεσημέρι για τις τροπολογίες σας. Μέχρι τότε μπορείτε να τις καταθέσετε. Ο Ιγνάτζιο Κουράου είναι εδώ, οπότε μπορούμε να πάμε στο σημείο 7 και να ξεκινήσουμε πιο νωρίς. Θα δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου και, της, και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Είναι μια έκθεση δική μας και έχει να κάνει με το κατά πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικές μας κατά πόσο συνεισφέρουν στις ε, παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε για αυτό το θέμα και το συζητήσαμε και πρόσφατα ε, στο πλαίσιο της ένδυσης ε, των, του ΦΛΕΚΤ και ο Ιγνάσιο έχει τώρα τον λόγο για να μας πει περισσότερα στοιχεία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, μάλλον έφτασα εγκαίρως. Όπως λέγατε, Πρόσφατα στο Κοινοβούλιο να γνωρίσαμε ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον σχετικά με τις επιχειρήσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εταιρική ευθύνη, ειδικά στον τομέα της ένδυσης, ε, τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, ε, τα ε, μεταλλεύματα που οδηγούν σε σειράξεις και το φλεκτ Οι πολιτικές ομάδες συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις ε, σε αυτά τα θέματα. Έχει ήδη ε, ψηφιστεί και εγκριθεί ένα σχέδιο με μεγάλη πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο. Ξέρουμε πολύ καλά λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για τον τομέα. δυστυχώ δεν έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον από την Κομισιόν. Οι βασικές ε, τροπολογίε έχουν κατατεθεί από διάφορες πολιτικές ομάδες, όμως έχουν κοινή κατεύθυνση από ό,τι φαίνεται. Ε, δεν υπάρχει μεγάλη απόκληση μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε όλες τις τροπολογίες σχεδόν στις συμβαστικές λύσεις. Έχουμε 22 συμβαστικές τροπολογίες. Ήδη υπάρχει δυνατότητα να κατατεθούν στις άλλες ομάδες και αύριο θα συναντηθούν οι σκιώδεις έτσι ώστε να οριστεί το κείμενο. Είμαι σίγουρος ότι το περιβάλλον εργασίας θα είναι ιδιαίτερα επικοδομητικό και το κείμενο που θα προκύψει θα είναι ξεκάθαρο και κοινή αποδοχής. Σε αυτό το ιδιαίτερα ε, θετικό κλίμα όμως θα κάνω ένα αρνητικό σχόλιο. Από τη μία το Κοινοβούλιο ε, έχει κοινή γραμμή για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Οι πολιτικές ομάδες έχουν το ίδιο όραμα, όμως από την άλλη η Κομισιόν συνεχίζει να αγνοεί τη φωνή μας συνεχώς ε, παρουσιάζει μια ριζικά διαφορετική ε, άποψη. Εδώ σε αυτή την επιτροπή και στην... έχουμε διαπιστώσει ότι στο DigiTrade υπάρχει διαφορετική προσέγγιση αντίθετα από αυτό που ζητά συνεχώς το Κοινοβούλιο. Τώρα για την εταιρική ευθύνη που έχει εγκριθεί τον περασμένο Οκτώβριο με μεγάλη πλειοψηφία δεν είδαμε κανένα follow-up από την Κομισιόν. Όταν ζητήσαμε απάντηση σε συγκεκριμένες ερωτήσεις πριν από μερικές ημέρες, η Κομισιόν ε, ε, έδωσε μια απάντηση που στην ουσία ε, είχε υπεκφυγές σχετικά με τα συγκεκριμένα πράγματα που ρωτούσε η συνεργασία με την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου θα μας βοηθήσει να θέσουμε και πάλι έμφαση σε κάποια ζητήματα που μας αφορούν και να ζητήσουμε την εφαρμογή του, των πραγμάτων που αποφασίσαμε τον Οκτώβρη. Με το Σκιώδης ε, θα ολοκληρώσουμε αυτό το έργο και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την συνεισφορά τους σε αυτή τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιο συνάδελφος να πάρει το λόγο. Μόνο η Χάιντι Χάουταλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Ιγνάσιο. Νομίζω ότι οι συμβαστικές σας λύσεις ε, θα είναι ιδιαίτερη ποιότητας. Δεν είμαι σκιώδης, όμως ήθελα να ρωτήσω εσάς και ίσως και την Κομισιόν κάτι, γιατί υπάρχει μια συνεχή συζήτηση για την εφαρμογή των ε, ε, ε, αρχών ε, ε, του Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και, την, και το επιχειρήν. Και υπάρχει και η διακυβερνητική πρωτοβουλία που εισήγαγε το Εκουαδόρ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω πώς σχετίζονται αυτές οι διαδικασίες μεταξύ τους. Η μία αποκλείει την άλλη, Πού είναι η έμφαση, το ρωτώ, γιατί ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κάποιες αμφιβολίες για αυτή την πρωτοβουλία του Εκουαδόρ και θεωρούσα ότι υπήρχε λόγος γι' αυτό, γιατί το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι η εφαρμογή. Αναφερθήκατε στο σχέδιο δράσης. Ε, τι γίνεται λοιπόν σε αυτό το τομέα. Τώρα μπαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τον κύριο Σένφελντ. Δεν υπήρξε σωστός χρονισμός, ζητώ συγγνώμη. Οπότε θα πρέπει να επαναλάβουμε τις ερωτήσεις εφόσον έρθουν σχετικά εγκαίρους. Κύριε Σένφελντ, θέλετε εσείς ε, μετά τους κοιότης να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αν κατάλαβα καλά, Πρόεδρε, συζητάμε για την αλυσίδα αυτή των αξιών, όπως είπατε. Μόλις μπήκα και δεν παρακολουθώ καλά. Πράγματι πρόκειται για την γνωμοδότηση πάνω ακριβώς στις σφαιρικές αυτές αλυσίδες αξιών. Περί αυτού πρόκειται και πάμε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι συνήθως. Ξέρω ότι δουλέψατε μαζί με τον Ινιάσιο Ευχαριστώ, λέει ο κύριο Ένφελτ. Ναι, μία ώρα νωρίτερα, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα παρόλα αυτά. Σχετικά με μένα, θα ήθελα να πω ότι αυτό το οποίο θα ήθελα είναι να ευχαριστήσω τον εισηγητή και αυτό γιατί το πρώτο σχέδιο γνωμοδότησης γύρω από το θέμα αυτό φαίνεται σωστό, ισορροπημένο. Λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση έτσι όπως επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις άλλες αγορές. Τα θέματα τα οποία επίσης μας απασχολούν μέσα στο έγγραφο αυτό είναι σημαντικά και για την ανάπτυξη και για την κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη είναι θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερος περίπλοκα. Είναι σαφές ότι είναι δύσκολο να αλλάξουν τα πράγματα γρήγορα και είναι δύσκολο να έρθουμε κοντά στις ευρωπαϊκές μας αξίες. Παρ' όλα αυτά ο εισηγητής νομίζω ότι καταφέρνει να αντικατοπτρίσει με τον σωστό τρόπο την σημερινή κατάσταση. Δεν συμφωνώ βέβαια με το 100% των προτάσεων και γι' αυτό έχω καταθέσει και έχουμε καταθέσει και γύρω στις 12 τροπολογίες, συνολικά 60 τροπολογίες έχουν κατατεθεί και 22 συμβιβαστικές. Ε, θα εξετάσω τις συμβιβαστικές, τις λάβαμε μόλις, αλλά βλέπω ότι πράγματι προσπαθούν να λάβουν υπόψη όλα τα σημαντικά σημεία και όλα τα ερωτηματικά τα οποία περιλαμβάνονται στις τροπολογίες τις μεμονωμένες. Έχει μεγάλη σημασία αυτό και αυτό που επίσης είναι σημαντικό στα πλαίσια της πρότασης που γίνεται στις συμβιβαστικές πρέπει ένα πράγμα να υπενθυμίζουμε συνεχώς ότι το κάθε κράτος είναι υπεύθυνο για τον σεβασμό του νόμου και εδώ καλείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει τον δικό της ρόλο. Δεν μπορούμε να είμαστε ε, ο αστυνομικός ε, του κόσμου όλου, δεν μπορούμε να δράσουμε έτσι, δεν χρειάζεται να παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά των άλλων. Δεν θα αντικαταστήσουμε εμείς τα κράτη-μέλη. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εξαγωγή γίνεται από τις χώρες και κάθε χώρα είναι υπεύθυνη γι' αυτά. Ο βασικός ρόλος λοιπόν των ευρωπαϊκών αρχών είναι να πιέσουν τις χώρες με τις οποίες έχουμε εμπορικές σχέσεις και οικονομικές σχέσεις, έτσι ώστε οι συγκεκριμένες αυτές χώρες να επιβάλλουν την τάξη στο έδαφος τους και να μην περιμένουν από μας να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτή ήταν η άποψή μου, την εξέφρασα και νομίζω ότι ελήφθη υπόψη και στις συμβιβαστικές. Ένα άλλο σημαντικό θέμα, τουλάχιστον για μένα σημαντικό, πρέπει να αναζητήσουμε κάποιες λύσεις οι οποίες να είναι δεοντολογικά σωστές μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτό είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνεται και στις συμβιβαστικές προτάσεις και με ικανοποιεί ιδιαίτερα. Ε, πρόσφατα ασχοληθήκαμε με το θέμα των ορυκτών. Είμαι πεπισμένος ότι τα πρότυπα τα οποία υιοθετήσαμε στα πλαίσια της έκθεσης για τα ορυκτά προϊόντα είναι ένα πρότυπο το οποίο θα μπορούσαμε να αναπαράγουμε εκεί όπου χρειάζεται. Υπάρχουν ε, α, συνάδελφοι με ιστορικού τύπου εμπειρίες εδώ, δουλέψαμε από κοινού, υπήρξε μια πλειοψηφία, την εγκρίναμε την πρόταση και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λογική αυτή και στο μέλλον. Λοιπόν, νομίζω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν και άλλοι που θέλουν το λόγο. Έιντι, ναι. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι η Κομισιόν θα εμφανιστεί για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον εισηγητή Ιγνάτσιο. Ναι. Πρώτα απ' όλα θα ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Βεβαίως και οι εισηγητές δεν είναι εδώ. Ε, σήμερα για τις τροπολογίες. Αύριο ελπίζω να βρούμε έναν καλό συμβιβασμό για το τελικό κείμενο που θα είναι αποδεκτό από όλους. Ε, η σχέση ανάμεσα ε, στις Έθνη, το Εκουαντόρ, αυτές οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι το πρόγραμμα εργασίας μας, είναι είναι ένα τομέα εργασία όπου θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μαζί κάτι καινούριο. Εάν από Ευρωπαϊκή πλευράς έχουμε μια πρόταση ε, καλή και γι' αυτό πρέπει να έχουμε την πρόταση και την συμμετοχή της Κομισιόν που δεν υπήρξε μέχρι τώρα με μια καλύτερη πρόταση, καλύτερους κανόνες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών και να μπορέσουμε ε, να συνεργαστούμε ε, για, με το Εκουαδόρ παραδείγματος χάρη, ε, με τον Ισημερινό, θα προσπαθούμε, μπορούμε να παίξουμε τον ρόλο μας ή τουλάχιστον να συμμετάσχουμε στο πλαίσιο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Αύριο θα έχουμε την συνεδρίαση με τους σκιώδεις συγητές και έχουμε 22 συμβιβαστικές τροπολογίες και θα δούμε ποιες θα είναι οι συμβιβαστικές τροπολογίες που θα λάβουν υπόψη τα σχόλια των συναδέλφων και θα ψηφίσουμε στις 3 Μαΐου. Συνάδελφοι, επειδή τώρα έχουμε ε, θα έχουμε κλείσει με, το, με την εργασία μας, ε, θα έχουμε την κίνηση συνάντηση ε, στην, κάτω στο, στην αίθουσα 3C στο ίδιο κτίριο με τις άλλες δύο επιτροπές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.